συναδέλφων, μπορώ να σας πω κύριε Μάιστατο ότι μπορείτε να βασιστείτε στην υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ευχαριστούμε πολύ. Έχει κλείσει η συζήτηση λοιπόν για την ετήσια έκθεση της ΕΤΕ για το 2009. Η ψηφοφορία θα γίνει σήμερα στις 12. Τώρα μπορούμε να περάσουμε στο επόμενο θέμα της ημερήσιας διάταξης που είναι η έκθεση του Γιάννους Βοητσικόφσκι Εμβολιασμό κατά του καταρροϊκού πυρετού του προβάτου» και δίνω το λόγο στον κύριο Βοητσικόφσκι. Ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, με μεγάλη μου χαρά θα σας παρουσιάσω την έκθεση αυτή για την τροποποίηση της Οδηγίας 2075 όσον αφορά τον εμβολιασμό κατά του καταρροϊκού πυρετού. Όπως ξέρετε, αυτή είναι μία ασθένεια που πλήττει τα μυρικαστικά της Ευρώπης και χαίρομαι διότι μερικά χρόνια πριν σας παρουσίασα την στρατηγική για την ευημερία των ζώων. Αυτό που κάνουμε σήμερα είναι ακριβώς αυτό. Μιλάμε για τον εμβολιασμό αυτό κατά του καταρροϊκού πυρετού και αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να προωθήσουμε τις δραστηριότητες για την πρόληψη αυτής της ασθένειας έτσι ώστε τα ζώα αυτά να βρίσκουν σε καλύτερη κατάσταση και η ασθένεια να μην σημαίνει ένα επιπρόσθετο κόστος. Η προηγούμενη οδηγία προσαρμόστηκε στις τότε συνθήκες και τα εμβόλια που τότε ήταν διαθέσιμα στην αγορά. Αυτά τα εμβόλια χρησιμοποιούνται και τώρα και βεβαίως υπό ορισμένους όρους. Γιατί αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να δούμε κατά πόσο ε, υπάρχει μεταδοτικότητα της ασθένειας με βάση τα παλαιά εμβόλια. Και αυτό που έχει σημασία είναι να λάβουμε υπόψη ορισμένες διαδικασίες, ότι θα πρέπει να εμβολιαστούν τα ζώα σε ένα συγκεκριμένο σημείο και ούτω καθεξής. Στο μεταξύ έχουν γίνει άλματα στην επιστήμη, έχουμε μία νέα γενεά εμβολίων έγιναν ε, οι κατάλληλες δοκιμές και αυτά τα νέα εμβόλια μπορούν πλέον να χρησιμοποιηθούν χωρίς να υπάρχει κανένας κίνδυνος ως προς τους προγενέστερους ε, περιορισμούς. Αυτά τα νέα εμβόλια θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν πολύ πιο εύκολα και αποτελεσματικά. E, αυτό που μας ενδιαφέρει λοιπόν είναι σε μικρό χρονικό διάστημα να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε και λάβαμε μία πρόταση νομοθετικού περιεχομένου από την Επιτροπή. Αυτό λοιπόν που μας ενδιαφέρει είναι να οργανώνονται οι εμβολιασμοί, να οργανωθούν φέτος το καλοκαίρι και γι' αυτό στις τροποποιήσεις και στις τροπολογίες της έκθεσης θέτω ορισμένες χρονικές προθεσμίες που θα πρέπει να αλλάξουν στις εθνικές νομοθεσίες για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις διατάξεις της οδηγίας για να μπορέσουμε να οργανώσουμε τους εμβολιασμούς φέτος και να μην περιμένουμε την παρέλευση ενός έτους. Υπάρχουν ορισμένα αμφιλεγόμενα σημεία βεβαίως. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε πίνακες συσχετισμού, ορισμένους ε, πίνακες συσχετισμού ή αντιπαραβολής. Και εμείς είπαμε ότι αυτοί οι πίνακες αντιπαραβολής θα πρέπει να υποβληθούν οι πίνακες συσχετισμού, οι αντιπαραβολής δείχνουν πώς αυτές οι διατάξεις έχουν μεταφερθεί στις εθνικές Ένωμες τάξεις. Ορισμένες, ε, ορισμένα κράτη το θεωρούν ως υπερβολική γραφειοκρατία. Αν όμως χρησιμοποιήσουμε αυτούς τους πίνακες αντιπαραβολής, έχουμε μια καλύτερη συνολική εικόνα για το τι συμβαίνει στα κράτη-μέλη και Συνεπώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτούς τους πίνακες για να πείσουμε τους πολίτες των κρατών μας γιατί συμβαίνει και ποια είναι η εξελικτική πορεία. Νομίζω ότι αυτοί οι πίνακες θα πρέπει να αποτελέσουν μια πάγια πρακτική στις νομοθετικές δραστηριότητες. Νομίζω ότι τώρα γίνεται κάτι το θετικό υπέρ των αγροτών και της ευζοίας των ζώων. Ευχαριστώ. Τώρα θα δώσω το λόγο στον κύριο Σέτκοβιτς, εξ ονόματος Ευρωπαϊκή Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ήθελα να ευχαριστήσει το Κοινοβούλιο για την στήριξη αυτή, στην στήριξη του μεγαλύτερου εμβολιασμού ε, κατά του καταρροϊκού πυρετού και θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον εισηγητή κύριο Βοχτσεκόφσκι για την στήριξη του. Ο καταρροϊκός έχει δημιουργήσει ιδιαίτερη ανησυχία στην κοινότητα των εκτροφέων στην Ευρωπαϊκή Ένωση από το, στην δεκαετία του 1990 θεωρήθηκε πως ήταν ε, μια εξωτική ασθένεια που σπάνια εμφανιζόταν στο νότο, αλλά τελευταία είχαμε κύματα επιδημιών σε αρκετά κράτη-μέλη και στην κεντρική και βόρεια Ευρώπη που δημιούργησαν μεγάλες απώλειες στο ζωικό κεφάλαιο αλλά και ε, αναταραχές στο εμπόριο ζώων. Έχει βελτιωθεί η κατάσταση με τον καταρροϊκό σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό σε μεγάλο βαθμό ε, χάρη στο μαζικό εμβολιασμό που συγχρηματοδότησε η Ευρωπαϊκή Ένωση. 150 εκατομμύρια ευρώ το 2008, 120 εκατομμύρια ευρώ το 2009 ε, και 100 εκατομμύρια ευρώ τα επόμενα χρόνια. Υπό τους τρέχοντες κανόνες εμβολιασμός επιτρέπεται μόνο στις περιπτώσεις όπου ε, υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί λόγω της ενδεμικής παρουσίας της ε, ασθένειας. Στην πρόταση εδώ της οδηγίας δίνουμε τη δυνατότητα να χρησιμοποιηθούν μη ενεργές ε, ουσίες για να εμβολιάσουν σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση έτσι ώστε να γίνει ένας προληπτικός ε, αδρανής με ένας προληπτικός εμβολιασμός ε, και σε περιοχές όπου δεν υπάρχει πρόβλημα για να μην φέρει το βάρος αυτό ο κλάδος ε, της γεωργίας. Είναι πολύ σημαντική η υγεία των ζώων και η ζωή των ζώων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και όντως επίγει το θέμα αυτό για να έχουν το χρόνο τα κράτη-μέλη ε, το χρόνο να εμβολιάσουν τα ζώα πριν ξεκινήσει η επόμενη περίοδος όπου ξεσπά ο καταρροϊκός. Παρόλο που έχει βελτιωθεί πολύ η κατάσταση τα τελευταία χρόνια δεν έχει εξαλειφθεί αυτή η ασθένεια και είμαστε πάντοτε υπό την απειλή νέων κυμάτων επιδημίας καταρροϊκού. Θα πρέπει λοιπόν να προστατεύσουμε τα ζώα από αυτό από αυτή την ασθένεια και θα πρέπει να μπορούν τα προγράμματα του εμβολιασμού να τα αυξήσουν ε, τα κράτη-μέλη ώστε να ανταποκριθούν σε μελλοντικέ επιδημίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάποια κράτη-μέλη ζήτησαν να εφαρμοστεί το μέτρο αυτό το συντομότερο δυνατό. Ο κύριος συγητής αναφέρθηκε στο πολύ δύσκολο θέμα των ε, πινάκων αντιπαραβολής, συσχετισμού που χρειάζονται για να δούμε αν μπορούμε να ε, διαπιστώσουμε το πώς έχει μεταφερθεί ε, πώς έχουν μεταφερθεί όλα αυτά τα μέτρα και οι προσπάθειες ε, που γίνονται στο εθνικό δίκαιο. Πώς μπορούμε λοιπόν τη μεταφορά των κοινοτικών διατάξεων να την εξασφαλίσουμε στο εθνικό δίκαιο μέσω αυτών των πινάκων. Έτσι μπορούμε να παρακολουθήσουμε ε, την σωστή μεταφορά του κοινοτικού δικαίου. Είμαστε απόλυτα σίγουροι πως με τέτοιου είδους επίγοντα θέματα και φακέλους όπως αυτό που συζητάμε σήμερα χρειαζόμαστε να δουλέψουμε σκληρά για να βρούμε μια λύση εδώ το Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και εμείς για να αποφύγουμε άχρηστα διέξοδα και εμπλοκές. Θέλουμε λοιπόν να έχουμε την απαραίτητη ευελιξία ώστε η νομοθεσία αυτή να εγκριθεί έγκαιρα και πρόθεσμα πριν ξεκινήσει πάλι η περίοδος όπως ξεσπάει ο καταρροϊκός πυρετός. Ευχαριστώ πολύ και τώρα θα ακούσουμε τις πολιτικές ομάδες. Η κυρία Γέγκλε, εξ ονόματος του ΕΛΚ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι. Η οδηγία την οποία συζητούμε σήμερα όσον αφορά τον καταραϊκό πυρετό είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα για την καταπολέμηση και την εξάλληψη αυτής της ασθένειας που πλήττει τα ζώα όχι μόνο τα πρόβατα εξάλλου αλλά και άρα μυρικαστικά, βοηδή. Το θέμα είναι ότι υπάρχουν διάφοροι τρόποι αντιμετώπισης ε, με εμβόλια αδρανοποιημένα, με εξασθενημένα ζώντα εμβόλια και με αυτόν τον τρόπο τα κράτη-μέλη μπορούν να χρησιμοποιήσουν με αποτελεσματικό τρόπο αυτόν τον εμβολιασμό έτσι ώστε να μειωθεί το βάρος που σήμερα πρίττει τον γεωργικό τομέα. Θα πρέπει να περιορίσουμε την ασθένεια αυτή και ελπίζω να δεχτούν τα κράτη-μέλη τις προδιαγραφές και τις ιδέες που προτείνονται. Αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα μια σημαντική βελτίωση της υγείας των ζώων. Όσο πιο ε, μαζικός είναι ο εμβολιασμός και πιο στοχευμένος περιοχές τόσο πιο μεγάλη θα είναι η αποτελεσματικότητά μας. Για να μπορέσει να ισχύσει αυτή η οδηγία και να είναι διαθέσιμα αυτά τα νέα εμβόλια, θα πρέπει να επιταχύνουμε τη διαδικασία. Η Αρμόδια Επιτροπή τη Δευτέρα στήριξε με μεγάλη πλειοψηφία αυτήν την ε, πρόταση και στηρίζω απόλυτα, όπως και η πολιτική μου ομάδα, την πρόταση του εισηγητή για τους πίνακες ε, συσχετισμού. Και αυτό θα πρέπει να γίνει διότι χρειαζόμαστε περισσότερη διαφάνεια και το λέω αυτό με πολύ συγκεκριμένο τρόπο στο Συμβούλιο. Τελειώνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την εξαιρετική του εργασία και για την εξαιρετική συνεργασία που είχε μαζί μας. Στηρίζουμε βεβαίως τις προτάσεις του. Ευχαριστώ πολύ κύριε Γέγκλε, λέει ο πρόεδρος. Βλέπω όμως τον κύριο Άγνιο που έχει μια ερώτηση. Τη δέχεστε? Έχετε το λόγο. Βάλτε όμως το μικρόφωνο σας ε, σε λειτουργία. Δεν είναι ερώτηση, είναι δήλωση. Δεν ήταν ομόφωνη η ε, υποστήριξη στην Επιτροπή. Ε, κύριε Άγνιου, όταν ε, χρησιμοποιείτε την μπλε κάρτα, να κάνετε ερώτηση. Χρησιμοποιείτε για ερώτηση. Και τώρα θα δώσω το λόγο στον κύριο Γκουτιέρες, εξ ονόματος των Σοσιαλιστών. Ευχαριστώ πολύ. Ο καταρροϊκός ε, πυρετός ήταν μόνη μια απειλή και για τα κοπάδια μας και για τη δημόσια υγεία. Ήταν μια ασθένεια την οποία προσπαθούσαμε να λύσουμε με το ζωντανό εμβόλιο έτσι ώστε να μην έχουμε περιορισμού στην κυκλοφορία των ζώων γιατί το πρόβλημα αυτό είναι ότι σε μη ε, μολυσμένα ζώα αν χρησιμοποιηθεί αυτό το μη αδρανοποιημένο εμβόλιο μπορεί να μεταδοθεί η ασθένεια. Αυτό δημιουργούσε λοιπόν πρόβλημα στο εμπόριο και για τους εκτροφείς γιατί είχαν να αντιμετωπίσουν τα αποτελέσματα της ασθένειας αλλά επίσης και επειδή περιοριζόταν η δυνατότητα ε, ε, εμπορίας των ζώων. Εάν έχουμε λοιπόν αυτό το αδρανοποιημένο εμβόλιο που επιτρέπει να μην έχουμε τέτοιου είδους αναταραχές στην ε, στην αγορά των ζώων, τότε θα πρέπει να το χρησιμοποιήσουμε για να καταπολεμήσουμε αυτή την ασθένεια. Όλα αυτά είναι ζωτική σημασία για ένα κλάδο. Άρα λοιπόν πρέπει να τροποποιήσουμε την οδηγία και να το κάνουμε το συντομότερο δυνατόν. Ξιότιμοι συνάδελφοι, η συμμόρφωση με τα όσα έχουμε στι συνθήκε και κυρίω με του πίνακε συσχετισμού δεν πρέπει να θεωρηθούν ω καλή δικαιολογία για να μην μπει σε εφαρμογή άμεσα η οδηγία γιατί η καθυστέρηση απλώ θα πλήξει ε, τους εκτροφείς. Η κυρία Πόλσον θα μιλήσει εξ ονόματος των ε, φιλελευθέρων και δημοκρατών για δύο λεπτά. Ευχαριστώ. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον κύριο Βοητσεκόφσκι για μια εξαιρετική εργασία. Ένα πολύ καλό κείμενο, πραγματικά. Οι συνάδελφοι ήδη είπαν περί τίνος πρόκειται. Πρόκειται για ένα νέο αποτελεσματικό εμβόλιο το οποίο να μπορέσει να χρησιμοποιηθεί σύντομα. Θα ήθελα λοιπόν στο λίγο χρόνο που διαθέτω να τονίσω το γεγονός ότι ίσως αυτό είναι το πρώτο αποδεικτικό απτό στοιχείο που δείχνει τι θα γίνει στο γεωργικό τομέα όταν αλλάξει το κλίμα. Στη Σουηδία, στη χώρα μου, μία ασθένεια ε, σαν αυτή του καταρροϊκού πυρετού ήταν κάτι το ανήκουστο μέχρι πέντε χρόνια πριν. Ήταν ε, μία σποραδική ασθένεια που βλέπαμε στο νότο της Ευρώπης. Τώρα όμως αποτελεί απτή πραγματικότητα και αντιμετωπίσαμε την πρώτη μας επιδημία πρόσφατα. Γι' αυτό θα πρέπει να αρχίσουμε με τον εμβολιασμό, αλλά επίσης θα πρέπει να κατανοούμε ότι όταν μιλάμε για το κλίμα, το περιβάλλον και τη μελλοντική τους εξέλιξη, να γνωρίζουμε ότι δεν πρόκειται για ξηρασία ή τροπικές βροχές. Εάν υποστούμε μείζονες κλιματικές αλλαγές, θα γνωρίσουμε μία εντελώς διαφορετική κατάσταση όταν πρόκειται για ασθένειες και επιδημίες και στα ζώα και στους ανθρώπους. Θα πρέπει λοιπόν να το λάβουμε υπόψη σοβαρά κατά τους υπολογισμούς μας όταν μιλάμε για την στρατηγική της Ευρώπης για το 2020. Επίσης, ως νομοθέτες, θα πρέπει να κατανοήσουμε ότι μπορούμε να λάβουμε σωστές αποφάσεις με βάση την παρούσα τεχνογνωσία και γνώση. Αλλά θα πρέπει να λάβουμε νέες αποφάσεις όταν ανακύπτουν νέα δεδομένα. Τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο στον κύριο Νίκολσον που θα μιλήσει εξ ονόματος των συντηρητικών και μεταρρυθμιστών. Ευχαριστώ. Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Βοτσεσκόφσκι για την έκθεση αυτή που συνέταξε και υπέβαλε στην Ολομέλεια. Εργάστηκε πολύ σκληρά. Θα ήθελα να μιλήσω για τους πίνακες συσχετισμού διότι ο Επίτροπος μας είπε ότι να είναι αρκετά καλή. Αλλά η ελπίδα δεν αρκεί, κύριε Επίτροπε. Είναι μια πολύ σοβαρή ασθένεια την οποία θα πρέπει να ελέγξουμε ήδη αυτό το καλοκαίρι. Γιατί τα μικρά αυτά έντομα μεταφέρουν την ασθένεια και θα πρέπει να την ελέγξουμε ήδη φέτος το καλοκαίρι. Ο κύριος Βοτσεσκόφσκι έκανε ό,τι μπορούσε και δεν μπορούμε να τον κατηγορήσουμε για οποιαδήποτε καθυστέρηση ή ολιγορία. Δυστυχώς στις Βρυξέλλες όμως υπάρχει μεγάλη γραφειοκρατία. Δεν πρέπει να ξεχνάμε όμως ότι η ασθένεια αυτή μεταδίδεται πολύ γρήγορα, ταξιδεύει πολύ γρήγορα και όπως είπε ο κύριος Βοτσεσκόφσκι και πολλοί άλλοι, η πρόληψη είναι καλύτερη από τη θεραπεία και νομίζω ότι θα πρέπει να κινηθούμε πολύ γρήγορα. Θα πρέπει να μας εξασφαλίσει η Επιτροπή ότι δεν θα υπάρξει περιττή γραφειοκρατία. Ο κύριος Άγνιου. Πρόκειται για μια ασθένεια όπου οι γεωργοί θα πρέπει να λάβουν τις δικές τους αποφάσεις ανάλογα με τις περιστάσεις. Εγώ από πλευρά των αγροτών του Ηνωμένου Βασιλείου δεν θα δεκτώ τη θέση των γραφειοκρατών. Ε, ε, θα πρέπει να σεβαστώ το Βρετανό φορολογούμενο. Εσείς μας δώσατε, μας μεταφέρατε αυτή την ασθένεια, μην επιδεινώνετε τα πράγματα. Το συζητάμε αυτό παρά τις εγγυήσει της συνθήκης της Λισαβόνας που δεν άλλαξε τα πράγματα. Γιατί λοιπόν αυτές οι αλλαγές θα πρέπει να επαναδιατυπωθούν για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν ξέρουμε πώς ε, θα επιληθεί το θέμα των πινάκων συσχετισμού και αυτό καταδεικνύει ε, τη σύγχυση που υπάρχουν στα πλαίσια της συναπόφασης. Ενώ η Βρετανική κυβέρνηση θα προσπαθήσει να δεχτεί τις ιδέες σας, αλλά κράτη-μέλη δεν θα τη δεχτούν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, και θα ήθελα να ευχαριστήσω και εγώ τον εισηγητή για αυτή την έκθεση. Γενικά τάσομαι υπέρ των αρχών που διέπουν αυτή την έκθεση, αλλά θα ήθελα να τονίσω ότι αυτός, αυτό το εμβόλιο θα πρέπει να δημιουργηθεί μόνο όταν οι αρμόδιες αρχές κρίνουν ότι υπάρχει κίνδυνος για το ζωικό κεφάλαιο στην Βόρειο Ιρλανδία και οι αγρότες και το Υπουργείο Γεωργίας εργάστηκαν πολύ σκληρά για να απαλλαγούμε από αυτή την ασθένεια. Θα πρέπει η Επιτροπή να δεχτεί αυτές τις ελεύθερες ζώνες και να ορίσει ε, ρήτρες περιφρούρησης. Όμως υπάρχει μεγάλος κίνδυνος διάδοσης αυτής της ασθένειας. Γι' αυτό θα πρέπει η Βόρεια Ιρλανδία να χρησιμοποιήσει, να μπορέσει να χρησιμοποιήσει τα ε, εμβόλια. Θα πρέπει οι αρμόδιες αρχές να εποπτεύσουν αυτό το εμπόριο και τις συναλλαγές έτσι ώστε να μην διαδοθεί η ασθένεια τα κράτη-μέλη θα πρέπει να καταγράψουν τους κινδύνους διάδοσης αυτής της ασθένειας και να προστατεύσουν την βιομηχανία για να μην υπάρξουν και άλλες αιστείες. Θα πρέπει λοιπόν να ελέγξουμε και να επιοπτεύσουμε αυτές τις αιστείες εκεί όπου υπάρχουν. Νικολέσκου. Ευχαριστώ οι επιδημίες όπως αυτή του καταρροϊκού πυρετού πλήττουν τους καταναλωτές και την ευρωπαϊκή οικονομία καθώς και την ε, θνησιμότητα των ζώων. Υπάρχουν πολλοί, περιορισμοί για την κυκλοφορία των, του ζωικού κεφαλαίου. Στα πλαίσια μιας εκστρατείας πρόληψης θα πρέπει να ορίσουμε ζώνες περιορισμού τη στιγμή που υπάρχουν ε, κρούσματα και πιστεύω ότι η πρόταση της Επιτροπής είναι ε, οικονομικά εύρωστη και πολύ σημαντική για τις μικρές εκμεταλλεύσεις. Επίσης, θα πρέπει τα ευρωπαϊκά ταμεία να βελτιώσουν την κατάσταση για τον περιορισμό του καταρροϊκού πυρετού. Έχει προωθεί Εκστρατείε μέσα στα πλαίσια 37 εκατομμυρίων τα τελευταία χρόνια θα πρέπει να υπάρξει κοινή χρηματοδότηση και τα επόμενα χρόνια έτσι ώστε να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε ε, μέσα στα πλαίσια της, των νομοθετικών ρυθμίσεων που ισχύουν μέχρι τώρα. Ευχαριστώ. Thank you. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Δεκάστρο. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω και εγώ τον κύριο Βοησεκόφσκι και όλους τους κοιόδης για αυτή την εργασία που καθιστά πιο ευέλικτες τις ρυθμίσεις για τον εμβολιασμό κατά του καταρροϊκού πυρετού. Καταβάλαμε κάθε προσπάθεια για να επιτρέψουμε αυτή την εκστρατεία εμβολιασμού πριν από το καλοκαίρι. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε υποβάλει μία πρόταση που δεν έλαμβανε υπόψη την έγκριση της συνθήκης της Λισαβόνας. Δηλαδή το Συμβούλιο έλαμβανε αποφάσεις χωρίς το Κοινοβούλιο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την νομική υπηρεσία του Κοινοβουλίου, διότι μπορέσαμε να αλλάξουμε τη νομική βάση δυνάμει του άρθρου 43 παράγραφος 2 της Συνθήκης μέσα στα πλαίσια της κοινή νομοθετικής διεργασίας. Τώρα περιμένουμε το Συμβούλιο με την ίδια αποτελεσματικότητα να δεχτεί τη θέση μας και τους πίνακες συσχετισμού έτσι ώστε να μπορέσουμε να δώσουμε μια άμεση απάντηση στις μικρές εκμεταλλεύσεις. Ο κύριος Έλουερντ έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Με την ε, χρήση αυτών των ε, εμβολίων και με τους περιορισμούς στην κυκλοφορία των ε, ζώων έχει μειωθεί ο επιπολασμός αυτής της ασθένειας τα τελευταία χρόνια. Έχει λοιπόν ένα πολύ μετρήσιμο αντίκτυπο στις κοινότητες υπαίθρου. Αυτό λοιπόν το αδρανές εμβόλιο σε περιοχές όπου δεν έχουμε σημειώσει κρούσματα αυτής της ασθένειας θα μας βοηθήσει πολύ. Μας δίνει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουμε τα πλέον εκτήματα που προσφέρει η παραγωγή αυτών των νέων τεχνολογίας εμβολίων και με τον τρόπο αυτό καταφέρνουμε να ξεπεράσουμε τα προβλήματα που είχαμε στο παρελθόν. Ο εμβολιασμός αποτελεί ένα αποδοτικό κτηνατικό μέτρο για τον καταρροϊκό πυρετό γιατί μπορούμε με τον τρόπο αυτό να εξαλείψουμε την ασθένεια στην Ευρώπη. Δηλαδή παρακολούθηση και εξάλληψη της ασθένειας θα πρέπει να αποτελέσουν τον απότερό μας στόχο και αυτό προς όφελος των Ευρωπαίων κτηνοτρόφων. Σας παρακαλώ πολύ να διαβάζετε πιο σιγά γιατί δεν προλαβαίνω διερμηνείς. Μα είναι περιορισμένος ο χρόνος μου κύριε Πρόεδρε. Η κυρία Γκέρλινγκ. Ευχαριστώ. Η νομοθεσία αυτή θα δώσει ευελιξία στους αγρότες και θα τους δώσει και ελπίδα, γιατί για πάρα πολύ καιρό η πολιτική εμβολιασμού παρεμποδίστηκε από το γεγονός πως δεν είχαμε αρκετά εξελιγμένα εμβόλια, έτσι ώστε να μπορούν να εμβολιαστούν τα ζώα εκτός ζώνων αποκλεισμού. Σε μια ζώνη αποκλεισμού, ε, μια ζώνη αποκλεισμού μπορεί να έχει τραγικά αποτελέσματα για τον κτηνοτρόφο και δεν προστατεύει και δεν προστατεύει τα ζώα τα ίδια από τις ασθένειες οι οποίες είναι πολλές φορές ε, εξαιρετικά ισχυρές όπως ο καταρροϊκός. Έτσι λοιπόν με τον εμβολιασμό θα επιτρέψει να εξαλειφθεί ο καταρροϊκός στο Ηνωμένο Βασίλειο, θα εξοικονομηθούν ε, χρήματα και θα σωθούν ε, ζωές. Θα πρέπει αυτοί οι κανόνες να τεθούν σε εφαρμογή το συντομότερο δυνατόν. Στις δυτικές περιοχές θα πρέπει να εμβολιάσουν πριν τα τέλη Μαΐου εκτινοτρόφοι έτσι ώστε να προστατευτούν απόλυτα τα ζώα από την ασθένεια. Όλοι κατανοούμε ποιο είναι το υπόβαθρο και τι είδους ε, μάχη έχει δοθεί για τους πίνακες σχετισμους στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά κτηνοτρόφια αυτά δεν τα καταλαβαίνουν και βασίζονται σε εμά ω ερετούς, ε, μια που είμαστε ερετοί του εκπρόσωποι για να τους βοηθήσουμε. Επίγει το θέμα και η κοινή λογική πρέπει να πρετανεύσει. α το ξεκινήσουμε και να κάνουμε μια επίγουσα διαδικασία fast track έτσι ώστε να εμβολιαστούν τα κοπάδια. Ευχαριστώ η κυρία Κέστιγκερ. Vielen Dank, Herr Präsident. Die Blauzungenkrankheit ist eine Tierseuche, die θα ήθελα να πω ότι πραγματικά τα πλήγματα από αυτή την ασθένεια είναι ήδη πολύ σημαντικά. Ήδη από το 2000 σε, σε πολλά κράτη-μέλη η επιδημία αυτή έχει πλήξει πολλά ζώα και πολλές περιοχές. Η οικονομική, αν θέλετε, πολύ αρνητική συνέπεια αυτής της ασθένειας είναι κάτι που απασχολεί πολλούς ε, γεωργούς. Θα πρέπει λοιπόν να βρούμε τρόπους να ανταπεξέλθουμε. Στην Αυστρία σε πολλές περιοχές έχει πλήξει η ασθένεια του καταρροϊκού πυρετού κοπάδια όχι μόνο προβάτων αλλά και βοηδών. Θα πρέπει λοιπόν εδώ να προσφέρουμε τη βοήθεια που χρειάζονται οι εκτροφείς μας γιατί ήδη από το 2000 η κατάσταση δεν, είναι, δεν αντιμετωπίζεται με ικανοποιητικό και αποτελεσματικό τρόπο. Σήμερα διαθέτουμε νέα εμβόλια, νέες τεχνολογίες και με πιο αποτελεσματικό τρόπο μπορούμε να μειώσουμε τα κρούσματα. Η χρησιμοποίηση αυτών των εμβολίων, των λεγόμενων ε, ζώντων εξασθενημένων, μας βοήθησε να περιορίσουμε ως ένα βαθμό σε κάποιες περιοχές την ασθένεια. Σήμερα όμως βλέπουμε ότι αυτό δεν αρκεί και πραγματικά θεωρώ ότι με πάρα πολύ ταχύ τρόπο θα πρέπει τα νέα μέσα που διαθέτουμε, τα νέα εμβόλια να χρησιμοποιηθούν στις περιοχές που πλήττονται ακόμα από την ασθένεια αυτή. Και αυτό θα πρέπει να γίνει πριν την νέα περίοδο, δηλαδή το νωρίτερο δυνατόν και αν είναι δυνατόν πριν τον Σεπτέμβριο. Ευχαριστούμε ιδιαίτερα τον εισηγητή. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Καπούλα Σάντος. Ευχαριστώ πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, οι προτάσεις σε, αυτή τη, σε αυτό το σχέδιο νομοθετικού περιεχομένου είναι πολύ καλές και χαιρόμαστε για την πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής λαμβάνοντα υπόψη και τις εξελίξεις της ε, επιστήμης έτσι ώστε να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε εμβόλια κατά του καταρροϊκού πυρετού πέρα από τις ζώνες αποκλεισμού έτσι ώστε να μην κυκλοφορήσει το μικρόβιο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον κύριο Βοητζεσκόφσκι της ε, Επιτροπής, από την Επιτροπή Γεωργίας καθώς και τη Νομική Επιτροπή για τη νομική βάση της πρότασης διότι όπως γνωρίζετε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι συνομοθέτη σύμφωνα με την ε, τακτική διαδικασία που εισήγαγε η συνθήκη της Λισαβόνας. Η Επιτροπή Γεωργίας ενέκνε την έκθεση σε σύντομο χρονικό διάστημα έτσι ώστε να γίνει ψηφοφορία σήμερα και να φτάσουμε στο επόμενο βήμα έτσι ώστε το Συμβούλιο να εγκρίνει και να μπορέσει να τεθεί σε ισχύ αυτή η οδηγία το ταχύτερο δυνατόν. Θα ήθελα λοιπόν το Συμβούλιο να λάβει υπόψη αυτές τις εξελίξεις γιατί είμαι σίγουρος ότι η έκθεση θα εγκριθεί με μεγάλη πλειοψηφία σήμερα. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, η νέα δυνατότητα εμβολιασμού για την καταπολέμηση της ασθένειας του καταρροϊκού πυρετού είναι κάτι που πραγματικά θα πρέπει να μας απασχολήσει. Η καλύτερη αντιμετώπιση είναι η πρόληψη. Και αυτό θα πρέπει να το σκεφτούμε και σε σχέση με αυτήν την οδηγία. Όλη αυτή η επιδημία μπόρεσε να περιοριστεί, αλλά τα πλήγματα συνεχίζουν να είναι πολύ σημαντικά. Οι περιοχές αυτές που έχουν πληγεί συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν προβλήματα. Εδώ λοιπόν και πολλά χρόνια αντιμετωπίζουμε μια πολιτική με μέσα τα οποία δεν αρκούν. Θεωρούμε λοιπόν ότι αυτή τη φορά πρόκειται για ένα πολύ θετικό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Θα ήθελα λοιπόν να αντιμετωπίσουμε το θέμα πιο συνολικά και άλλα ζώα πλήττονται σήμερα και η κλιματική αλλαγή μας οδηγεί σε μια πολύ πιο γενική ε, αντιμετώπιση. Θεωρώ ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορεί συνέχεια να καθυστερεί και να συζητά θέματα τα οποία φαίνονται σήμερα ότι είναι η μόνη λύση. Στηρίξαμε την έρευνα, στηρίξαμε τις νέες τεχνολογίες και θεωρούμε ότι μια επικίνδυνη ασθένεια μπορεί σήμερα να αντιμετωπιστεί. Έχουμε μια νέα κατάσταση. Ευχαριστώ ιδιαίτερα τον εισηγητή, ο οποίος με μεγάλη ταχύτητα προετοίμασε την έκθεσή του και ελπίζω ότι θα είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση, να βοηθήσουμε τα κράτη-μέλη να μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν και να διαθέσουν στους εκτροφείς αυτά τα νέα εμβόλια. Πρόκειται για πιο αποτελεσματικά εμβόλια τα οποία κατά την άποψή μου θα πρέπει το ταχύτερο δυνατόν να είναι διαθέσιμα. Βεβαίως η Επιτροπή σήμερα βλέπουμε ότι θα πρέπει να επεξεργαστεί καλύτερα τις προτάσεις. Θα πρέπει να προσαρμοστεί στις νέες διαδικασίες και αυτό με μεγάλη ταχύτητα. Όσο γρήγορα δουλεύουμε εδώ στο Κοινοβούλιο θα πρέπει να δουλέψει και η Επιτροπή. Γιατί αλλιώς η νέα αυτή τεχνολογική πρόοδος δεν θα μπορέσει εγκαίρως να χρησιμοποιηθεί. Θέλετε παρέμβετε στην ε, ε, παρέμβαση, να μιλήσετε επί της ε, παρέμβασης του Νέλ Χάρτ. Όχι, για το Catch Day. Εντάξει, ο κύριος Ταραμπέλα έχει το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Γιάννου και για την έκθεσή του που μας υπενθυμίζει πόσο σημαντική είναι η νομοθεσία που έχει προσαρισμεί. Το κατά πόσο θα είναι αδρανές ή όχι το εμβόλιο τι να σας πω, στις αναλύσεις αίματος δεν είναι εύκολο να εντοπιστεί και να απομονωθεί είτε στο ζώο ε, εάν αυτό είναι ήμερο είτε αν όχι να απομονωθεί και να βρεθεί εύκολα στο αίμα του. Άρα λοιπόν καλό θα είναι να δούμε πώς μπορούμε να κάνουμε τη διάκριση μεταξύ ενός εμβολιασμένου ε, ζώου και ενός ζώου που έχει προσβληθεί. Γιατί ο κίνδυνος με ένα προσβεβλημένο ζώο είναι ιδιαίτερα μεγάλος και είδατε τι γίνεται, ε, για παράδειγμα με τις χώρες που ήδη χρησιμοποιούν το αδρανές εμβόλιο. Θα πρέπει λοιπόν εμείς να βρούμε μια, ένα εμβόλιο το οποίο θα δίνει μεγαλύτερη βιοασφάλεια έτσι ώστε να δώσουμε μια καλύτερη υγειονομική και εμπορική απόκριση στο θέμα αυτό το οποίο είναι τόσο δύσκολο. Τώρα φτάσαμε στο διαδικασία της αυθόρμητης παρέμβασης, στο Catch the Eye. Κυρία Μαγκίνης είναι η πρώτη ομιλήτρια. Ευχαριστώ πολύ. Καλό θα ήταν να υπενθυμίσουμε τα όσα είπε ο Επίτροπος, δηλαδή έχουμε, έχουν μειωθεί τα κρούσματα σε 120 το 2010 από 40.000 πριν από 4 χρόνια. Τώρα θα πρέπει να δούμε τι γίνεται με το δρανέ εμβόλιο και με την χρήση του και τις τεχνικές λεπτομέρειες. Αυτό θα ήταν ιδιαίτερα καλοδεχούμενο. Εάν λοιπόν ήταν εδώ το Συμβούλιο, θα μπορούσαμε να συζητήσουμε το κατά πόσο υπάρχει η βούληση να παρουσιάσουμε τους πίνακες συσχετισμού που θεωρούν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Κοινοβούλιο όπως είναι απαραίτητοι. Και θα ήθελα να έχουμε μια απάντηση πολύ σύντομα για το θέμα αυτό. Πρόληψη ασθενειών, πολύ σημαντικό αλλά αυτό έχει να κάνει επίσης ε, και με τον πολλαπλασιασμό των ζώων και με τους ξενιστές, του φορείς και όλα τα θέματα τα οποία ε, συζήτησαμε σήμερα το πρωί. Οπότε υπάρχει το θέμα αυτό με το εμβόλιο. Ευχαριστώ πολύ. Κύριος Λάσα έχει ζητήσει το λόγο. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να σας ε, αναφέρω το εξής, ότι σε ουρολογικές, ε, ορολογικές έγινες που έρευναν, έρευνες που έγιναν ελέγχθηκε το κατά πόσον τα ζώα είναι πράγματι ασθενή. Ε, για να διαπιστωθούν λοιπόν τα τελικά αποτελέσματα θα πρέπει όπως σας είπα να γίνουν αυτές οι ορολογικές εξετάσεις και αυτό δημιουργεί πρόβλημα στη μεταφορά των ζώων. Κυρίως διότι εκείνο που ενδιαφέρει είναι η μεταφορά της οδηγίας στην νομοθεσία των κρατών μελών. Και αυτό είναι αδύνατο να επιτευχθεί το 2011. Εγώ προσωπικά δεν συμφωνώ με αυτήν την ομοιρία, δηλαδή την 20η ημέρα και θεωρώ ότι αυτή η προθεσμία πρέπει να παραταθεί. Πρέπει να έχουμε κατά νου ότι οι κατάλογοι που θα επεξεργαστούμε θα οδηγήσουν σε αύξηση του διοικητικού κόστους. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι πρόκειται για ένα βήμα προς τα εμπρός για να κατανοήσουμε ότι δεν είναι ένα θέμα που αφορά ορισμένες ε, ε, περιοχές ε, βορείως της Αφρικής, δηλαδή στη Νότια Ευρώπη. Εν πάση περιπτώσει θεωρώ ότι η διάταξη είναι πολύ καλή και θα ήθελα να υποβάλω ένα ερώτημα προς τον κύριο Ταραπέλα. Δεν θεωρεί η Επιτροπή, ο συνάδελφος, ότι θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε άμεσα και το θέμα της εφαρμογής στις ε, κτηνιατρικές υπηρεσίες, διότι ίσως να μπορέσουμε να εξαλείψουμε το πρόβλημα, την ασθένεια σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο κύριος Γιάρ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ε, το να υπάρχουν καλύτερε συνθήκε εμβολιασμού για την αντιμετώπιση αυτή τη ασθένεια είναι πολύ σημαντικό γιατί μόνο με το ενεργό εμβόλιο μπορούν οι παραγωγοί να αντιμετωπίσουν τον κίνδυνο ε, περαιτέρω μόλυνσης. Θα πρέπει λοιπόν ε, να μεριμνήσουμε έτσι ώστε να μην εμφανιστεί και ο αυθόδης πυρετός. Πρέπει να έχουμε επίσης κατά νου ότι η γεωργία είναι ένας ε, σημαντικός τομέας ε, για όλα τα ευρωπαϊκά κράτη-μέλη και κατόπιν τούτου οι γεωργοί πρέπει να έχουν στα χέρια τους τα πιο σύγχρονα ε, ιατρικά πορίσματα για να μπορούν να εκμεταλλευτούν σωστά αυτά που προσφέρουν τα εμβόλια. Αυτά λοιπόν που χρειαζόμαστε είναι δύο πράγματα. Πρώτον, χρειαζόμαστε μια ταχεία λύση η οποία να εφαρμοστεί στην πράξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και δεύτερον, χρειαζόμαστε εξίσου επιγόντως ε, της, ε, τη δήλωση και την ανακοίνωση από πλευράς Κομισιόν στα κράτη-μέλη ότι είναι υποχρεωτικό να τις ανακοινώνουν τις περιπτώσεις που προκύπτουν. Και τέλος ο Επίτροπος έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ξεκινήσω ευχαριστώντας το Κοινοβούλιο για την τεράστια στήριξη αυτής της πρότασης, όπως επίσης και για το ότι αναγνωρίσατε πως το θέμα αυτό επήγε και πως χρειαζόμαστε διαδικασίες ταχύτατες. Αναφερθήκατε στο πρόβλημα των πινάκων συσχετισμού και θα ήθελα να σας υπενθυμίσω πως το θέμα αυτό το έθεσε και η διάσκεψη των ε, Προέδρων η οποία προσπάθησε να μας κινητοποιήσει στο σημείο αυτό μια και βλέπει πως το θέμα της μεταφοράς ευρωπαϊκής νομοθεσίας στο, στην εθνική νομοθεσία εξακολουθεί να υπάρχει. Είναι τόσο δύσκολο άραγε mm. να κοινοποιεί κανείς ως κράτος μέλος ε, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ποια τμήματα της ευρωπαϊκής νομοθεσίας έχουν μεταφερθεί και με ποιο τρόπο. Είναι τόσο δύσκολο γιατί τη στιγμή που ανασχολούνται με το πώς θα γίνει αυτή η μεταφορά, φαντάζομαι πω κάνουν κάποιες πως κανουν καποιε προσπαθειες προετοιμασια και λαμβάνουν κάποιε αποφάσεις για τη μεταφορά αυτή. Άρα λοιπόν αναγνωρίζουμε όλοι και ακούστηκαν αρκετές συζητήσει στο σημείο αυτό για το πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση υποφέρει όταν η μεταφορά της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας γίνεται με άνισο τρόπο. Επειδή λοιπόν το έχουμε συζητήσει για τη συγκεκριμένη νομοθεσία ενδεχομένως να είναι και βλαβερή η ελληπής η καθυστερημένη μεταφορά. Όπως είπα και στα αρχικά μου σχόλια και επαναλαμβάνω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι σαφώς κατά των α, μη απαραίτητων εμπλοκών. Ναι, επήγε το θέμα. Θέλουμε μεγαλύτερη ευελιξία. Θέλουμε να γίνουν εντατικέ διαπραγματεύσεις έτσι ώστε να βρεθεί μια λύση. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα προσπαθήσει να είναι όσο κρίσιμη μπορεί να σας φανεί. Μια και πρέπει να ξεκινήσει ο εμβολιασμό πριν ξεκινήσει η περίοδος επιπολασμού της ασθένειας. Τώρα για το κατά πόσο είναι έτοιμη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εφαρμόσει τα μέτρα αυτά, θα ήθελα ε, τον κύριο Γκέρ και τον κύριο Σελχάρη να τους εξασφαλίσω όπω κάναμε ό,τι μπορούσαμε και τα εφαρμοστικά μέτρα είναι σχεδόν έτοιμα. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι η έγκριση. Έγκριση των προτάσεων αυτών από τον νομοθέτη. Αφού κλείσει αυτό θα προχωρήσουμε με πολύ ταχύ ρυθμό. Σας ευχαριστώ και πάλι, ευχαριστώ τον εισηγητή και σα ευχαριστώ για την πολύ άριθμη στήριξη που προσφέρατε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ ε, για όλα αυτά που είπατε, που με στηρίξατε. Επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους εσκαιώδης ηγητές και τα μέλη της Επιτροπής Γεωργίας. Σας ευχαριστώ πολύ που μας επιτρέψατε να εργαστούμε τόσο γρήγορα. Είναι σπάνιο στο Κοινοβούλιο να μπορούμε να εγκρίνουμε έγγραφα τα οποία συνεπάγονται βελτίωση της κατάστασης των πραγμάτων. Νομίζω ότι είναι δύσκολο για μας ε, να κατανοήσουμε και να αισθανθούμε συμπάθεια για την οποιαδήποτε εθνική γραφειοκρατία. Δεν είναι τόσο δύσκολο να ε, προετοιμάσουν τα στοιχεία και να τα στείλουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Από την άλλη όμως ε, είναι πολύ πιο δύσκολο για έναν απλό πολίτη να γνωρίζει κατά πόσον η ε, νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει μεταφερθεί στη δική του τη χώρα ή όχι. Έτσι λοιπόν αυτοί οι πίνακες αντιστοιχίας θα είναι χρήσιμη για όλους μας και θα είναι ένα πραγματικά χρήσιμο έγγραφο. Ε, απευθύνομαι λοιπόν ε, σε εσά ε, στο ε, Συμβούλιο ε, να μην κάνετε αυτόν τον αγώνα απαραίτητα, να μην διαφωνήσετε με αυτούς τους πίνακες αντιστοιχία. Ας ελπίσουμε ότι φέτος το καλοκαίρι θα διεξάγουμε αυτή την εκστρατεία για τον εμβολιασμό γιατί αλλιώς αν δεν γίνει κάτι τέτοιο θα είναι τζάπα η δουλειά μας. Δεν θα έχει οδηγήσει σε τίποτα. Πολύ ωραία λέει ο Πρόεδρος. Ε, ολοκληρώθηκαν οι εργασίες μας για το θέμα αυτό. Θα ψηφίσουμε στις 12 και ε, το επόμενο θέμα είναι κοινοτικές εισαγωγές τομάτας από το Μαρόκο. Πρώτη μιλήτρια η κυρία Ματσόνη.